Er- Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίασή μας. Έχετε την ημερήσια διάταξη στα χέρια σας. Έχετε παρατηρήσεις ή κάποιες επιθυμίες αλλαγών. Δεν υπάρχουν. Τότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο ημερήσιας διάταξης. Είναι η έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης. Πάντα μέχρι τέλος της συνεδρίασης, μέχρι της συνεδρίασης, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρείται πάντα ότι κυρώνονται, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και μετά ανακοινώσεις Προέδρου. Ως εξής έχουν οι ανακοινώσεις Προέδρου. Θέλω να υπενθυμίσω αφενός ότι και αυτή η συνεδρίαση ζωντανά στο διαδίκτυο μπορεί να παρακολουθείτε και να το σκεφτείτε μπορεί κάποιος να σας δει απ' έξω να φέρεστε λοιπόν με τον δέοντα τρόπο έχουμε και ένα κατάλογο μια κατάσταση των, της αλληλογραφίας και αν σας ενδιαφέρει μπορείτε από τη γραμματεία να ζητήσετε αντίγραφο έχουμε και μια επίσημη είχαμε μια επίσημη συνεδρίαση με την TPC την Επιτροπή Εμπορίου του Συμβουλίου που συνεδριάζει την Παρασκευή και ανταλλάξαμε απόψεις ε, για την πολιτική γενικότερα, για το εμπόριο και για το θέμα των TDIs και IPIs, των σημαντικών δηλαδή νομοθετικών διαδικασιών. Ωστόσο όμως με μικρή πρόοδο. Σίγουρα αύριο θα το ξαναδούμε με την Ιταλική Προεδρία, υφυπουργό εμπορίου της Ιταλίας, της Προεδρίας του Συμβουλίου, που έχει την ε, ευθύνη για τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο. Φιλοξενήθηκα και από την επίσημη συνεδρίαση Υπουργών Εμπορίου 21 Νοεμβρίου. Και λέω ότι δεν είναι κάτι το μοναδικό αυτό ως προηγούμενο, αλλά ως θέμα αρχής θα συναντώμεθα με τους αρμόδιους υπουργούς σε τακτά διαστήματα και για τις διαπραγματεύσεις για την TTIP όσον αφορά την Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τις ΗΠΑ αλλά και τα TDI τα μέσα της άμυνας αλλά είναι ενδιαφέρουσα και η συζήτηση με την Κίνα δεδομένων των οικονομικών προκλήσεων αλλά και λόγω των νομικών προβλημάτων που απορρέουν σε σχέση με το εμπόριο με την Κίνα. Μετά, ύστερα ήθελα να σας ενημερώσω ότι του χρόνου 2015 οι τροπολογίες δεν θα υπογράφονται προσωπικά, δεν θα είναι υποχρεωτικό αυτό. Ηλεκτρονικά θα μπορούν να υπογράφονται, να προσυπογράφονται στη νέα πύλη, διαδικτυακή πύλη Signal Portal, Digital Signal Portal, ψηφιακή δηλαδή ε, πύλη του διαδικτύου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό το μέσο, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά. Έπειτα θέλω να χαιρετήσω θερμά να τον καλωσορίσω τον Μακ που βρίσκεται δεξιά δίπλα στον Αλμπέρτο. Είναι νέος ε, όσον αφορά τη γραμματεία της Επιτροπής μας αντικαθιστά τον Νίκολας Ντοζρέτ που αποχώρησε και πήγε σε άλλη θέση διοικητική. Χαιρόμαστε, για, προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία και ευχόμαστε, ελπίζουμε να αισθάνεσαι σπίτι σου. Στο τέλος της συνεδρίασης σήμερα θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί είναι η τελευταία περίοδος συναντήσεων πριν από την ε, αλλαγή της χρονιάς Μπορούμε στο τέλος να προσκαλέσουμε λοιπόν σε μια συνάντηση κατά το τέλος όμως της συνεδρίασης μπροστά στην αίθουσα θα γίνει αυτό και μετά να επισημάνω ότι στο πλαίσιο του ΠΟΕ Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ευτυχώς σημειώθηκαν σημαντικές σαφείς πρόοδοι μια και τα προβλήματα όσον αφορά την Ινδία για παράδειγμα και προγράμματα ασφάλειας τροφίμων προσωρινά επιλήθηκαν και είχαμε την έγκριση των trade facilities των διευκολύνσεων εμπορίου του Μπαλί. Και φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά το γύρο Ντόχα και έχουν, μπορούν να πάρουν πάλι να δρομολογηθούν. Και είναι ένα σημαντικό σημείο και αυτό, διότι στο σημείο των κυριότερων σημείων που θα συζητηθούν στη μελλοντική εμπορική πολιτική πρέπει αυτά να ληφθούν υπόψη. Χθες το βράδυ στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χθες το βράδυ, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου συνήλθαν με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν επαφές, συζητήσεις. Και σε αυτές τις συζητήσεις επρόκειτο φυσικά για τα 10 κέντρα βάρους της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ένα από τα δέκα αυτά κέντρα βάρους είναι η έγκριση ενός δίκαιου και ισότιμου πλαισίου συμφωνίας εμπορικής με τις ίπα. Ορθό και σημαντικό αυτό, αλλά δεδομένης της εξέλιξης που υπάρχει σε σχέση με τον ΠΟΕ, είναι πάρα πολύ σημαντικό τις πολυμερείς πτυχές του εμπορίου να μην τις αμελήσουμε, να μην τις αγνοήσουμε και όσον αφορά την διαδικασία του ΠΟΕΚ και αυτή να θεωρηθεί κέντρο βάρος και έτσι να την προσέξουμε. Το ανέφερα αυτό και χθες το βράδυ επιπρόσθετα. Πολύ καλά. Λοιπόν, δεν ολοκληρώσα, δεν τέλειωσα. Περνάω τώρα στο θέμα της διαφάνειας. Δηλαδή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Αρκετό χρονικό διάστημα είχαμε διαφορές σε σχέση με την προσπάθεια δημιουργίας περισσότερης, μεγαλύτερης διαφάνειας. Το συζητήσαμε και με επιτρόπους, αλλά και πέρα από αυτό υπήρξε αντίδραση από την αρμόδια επίτροπο και η πρόταση για μια πρωτοβουλία για τη διαφάνεια υποβλήθηκε, κατατέθηκε, πράγμα που το χαιρετίζω. Τώρα εξειδικευμένα, πιο καταλεπτός θα πρέπει να προχωρήσουμε στη δουλειά στο συγκεκριμένο έργο και αυτό δεν είναι τόσο απλό διότι φυσικά υπάρχουν σημαντικά διοικητικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή το ότι τέτοιου είδους έγγραφα για 751 βουλευτές που πρέπει να διανέμονται και δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση και σε σχέση με τη γραμματεία μας εδώ οι συνάδελφοι σχεδόν θα είναι αποκλειστικά απασχολημένοι μόνο με εμπιστευτική ανταλλαγή και διαβίβαση εμπιστευτικών εγγράφων. Μεγάλη επιβάρυνση. Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρωτοβουλία για απλούστευση και διαφάνεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Και τέλος η ανακοίνωση Προέδρου σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά το περιβάλλον και τα αγαθά. Είχαμε το δεύτερο γύρο όσον αφορά το Σεπτέμβριο και είχαμε τον διορισμό, τον καθορισμό ε, αυτών των ε, αγαθών και μετά παράλληλα με την ε, συνεδρίαση έχουμε τον κατάλογο αυτών των προϊόντων που θα συζητήσουμε, θα συζητηθεί ιδιαίτερα όσον αφορά την οδηγία για το, για το νερό ε, και ε, την ποιότητά του. Τέταρτος γύρος προβλέπεται για τον Ιανουάριο 2015 και τα 14 μέχρι σήμερα μέλη ενισχύθηκαν. Η Ισλανδία είναι τώρα και εκείνη μέρος των διαπραγματεύσεων προσθέθηκε και εκείνη στην ομάδα των διαπραγματευτών. Αυτό είναι μια καλή προσέγγιση όσον αφορά τις προσπάθειες του ΠΟΕ. Πολύ καλά, περνάμε στο σημείο 4. Είναι το θέμα των τριμερών διαλόγων αυτό. Έχουμε να αναφέρουμε μόνο για ένα τριμερή διάλογο που ολοκληρώθηκε, έγινε με το Συμβούλιο. Ε, πρόκειται για το νομοθετικό έργο για τα εξωτερικά εμπορικά στατιστικά στοιχεία. Πράγμα που με μια πρώτη ματιά δεν φαίνεται τόσο πολιτικά ευαίσθητο ή φλέγον θέμα, όμως τεχνικά και διαδικαστικά και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ερώτημα, το ζήτημα είναι ποια στοιχεία της νομοθεσίας στο βασικό κείμενο μπορούν να ενταχθούν. Ποια θα ε, ε, ενταχθούν σε ένα πλαίσιο κατεξουσιοδότηση πράξεων και η δική μας θέση φυσικά είναι ότι όλα εκείνα τα οποία αφορούν ρυθμιστικές προτάσεις θα πρέπει να βρίσκονται είτε στο βασικό κείμενο είτε σε μια κατεξουσιοδότηση πράξη. Όχι όμως σε μια εφαρμοστική ε, πράξη ή οδηγία. Κατά τούτο λοιπόν σε αυτόν τον τρίλογο, τριμερή διάλογο, πρόκειται για αυτό το θεσμικό θέμα. Την επόμενη Δευτέρα στις 8 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια νέα συνάντηση για αυτό το ζήτημα. Και μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στα επίμαχα θέματα να υποβάλει συμβιβαστικές προτάσεις. Χαρακτηρίστηκε ο πρώτος γύρος συζητήσεων από την επιθυμία να υπάρξει συμφωνία. Και η Ιταλική φυσικά Προεδρία του Συμβουλίου θα διαδραματίσει πολύ επικοδομητικό ρόλο, είναι βέβαιο. Και έτσι υποθέτω και λέω ότι αυτό το πνεύμα, το συμβιβαστικό πνεύμα την επόμενη Δευτέρα θα χαρακτηρίσει τις διαπραγματεύσεις για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε πολύ καλά. Δεν ζήτησε κανείς τον λόγο και έτσι μπορούμε πολύ καλά. Πήγαμε πολύ γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Είχαμε επιταχύνει. Δεν βρίσκεται εδώ με. Έστω, δεν πειράζει. Θα προτείνω να αλλάξουμε τη σειρά. Και να περάσουμε στο σημείο 6 για να μην υπάρξει κενό χρονικό διάστημα. Το 6 τι είναι, είναι η απαλλαγή 2013. Και δίνω τον λόγο για αυτό το θέμα στον αξιότιμο και ικανότατο εισηγητή για τον προϋπολογισμό Ράιμερ Μπέγκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Ευχαρίστως να το κάνω λοιπόν. Αλλά ε, φυσικά μπορεί, να υπάρχει ε, ίσως η απέτηση να ε, ομιλώ μέχρι να έρθει το ελεκτικό συνέδριο, δύσκολη υπόθεση και για τις γενικές προτιμησιακές ρυθμίσεις και ένα ουσιώδες στοιχείο της δικής μας γνωμοδότησης για τη χορήγηση απαλλαγής θα πρέπει θέματα να συζητηθούν, χωρίς να προδικάσω τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο, αξίζει να δει κανείς αυτή την ε, περίληψη. Διότι με το παράδειγμα των προτιμησιακών ε, εμπορικών συμφωνιών και το ζήτημα που βρίσκονται τα πιο αδύναμα σημεία, ευάλωτα σημεία, είναι υπόδειγμα αυτό για να δούμε κάποια άλλα θέματα του προϋπολογισμού. Το ένα είναι ποια είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποια ευάλωτα σημεία υπάρχουν εκεί σε σχέση με αυτό το θέμα. Πού υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών και ποιες ρυθμίσεις, ποια μέρη να λαμβάνεται ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα ευαίσθητα, ευάλωτα θέματα. Να πω όμως το εξής για τη χορήγηση απαλλαγής. Μόνιμα έχουμε αυτή την δημόσια συζήτηση για τη δήλωση ε, αξιοπιστίας, δηλαδή η δήλωση, η βεβαίωση αξιοπιστίας του ελεκτικού συνεδρίου που καμιά φορά δημιουργεί κάποια προβλήματα. Δυστυχώς όμως στην πολιτική δημόσια συζήτηση τι συμβαίνει. Όλα τα ρίχνουμε σε ένα καζάνι. Ισοπεδωτικά τα αντιμετωπίζουμε. Θυμάμαι κάποια συζήτηση που είχαμε στις Βρυξέλλες με τον, την τότε αντιπρόεδρο Χέντα Φαρβέντερ που ήταν και πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Γερμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου σε μια συζήτηση που ήταν πολύ επίμαχη είπε το εξή. αν είπε τα κράτη-μέλη ένα τέτοιο σύστημα όπως τη δήλωση αξιοπιστίας υπόκειντο σε αυτήν τότε η πλειοψηφία των κρατών μελών μια τέτοια δήλωση δεν θα την έπαιρναν μια τέτοια δήλωση αξιοπιστίας από το ε, ελεκτικό συνέδριο. Αυτό για να αποσαφηνίσουμε πετίνος πρόκειται. Και μετά για το ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου. Πού βρίσκονται τα ουσιοδέστερα προβλήματα που έχουμε για την ε, διεκδίκηση ή απέτηση βέλτιστης χρήσης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά γνωρίζουμε ότι μεγάλα τμήματα του προϋπολογισμού τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα όχι μόνο το εθνικό επίπεδο έχουμε αλλά και το περιφερειακό επίπεδο για την υλοποίηση της κοινή αγροτικής πολιτικής ή των διαθροτικών πολιτικών της Ένωσης π.χ. Να δώσω μια επισήμανση. Επί χρόνια στην Επιτροπή Προϋπολογισμών διαπραγματευόμασταν και λέγαμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών θα πρέπει μια εγγύηση να μπορούν να, να συντάξουν για τη σωστή χρήση και διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επί χρόνια το υπονόμευαν αυτό ως πρόταση. Σημαντικά κρατημέλη κιόλα. Επειδή υπάρχουν λέει ομοσπονδιακές δομές, δεν μπορεί ο ομοσπονδιακός υπουργό να διασφαλίζει το τι γίνεται σε κάθε κρατήδιο. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με τα όσα αναμένονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορεί να γίνει στα κρατημέλη. Τι δείχνει αυτό. Αυτό δείχνει ότι ο Μουντζούρης περνάει σε άλλα χέρια και κατηγορούνται κάποιοι για τέτοιες καταστάσεις. Παρόλα αυτά είναι σαφές ότι σε κάποια χρήση, κάποιες χρήσεις κονδυλίων, ευρωπαϊκών κονδυλίων, το ζήτημα της ευρωπαϊκής πρόσθετης αξίας ή το θέμα των επιπτώσεων πιθανώς δεν ελέγχεται επαρκώς. Είμαι ευγνώμων στο ελεκτικό συνέδριο για το ότι κατά τα τελευταία χρόνια λίγο πιο σε βάθος ε, επεξηγεί ότι ο περίπλοκος χαρακτήρας ε, Τέτοιου είδους ρυθμίσεις για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα του ζητήματος. Οι πολίτες το θεωρούν απάτη αυτό εντός εισαγωγικών, περιπτώσεις απατών. Όμως υπάρχουν επιπτώσεις λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα ρυθμίσεων και διατάξεων που ξεπερνούν πολλές φορές την ε, δυνατότητα των ε, απλών ανθρώπων να ανταπεξέλθουν. Και είναι θέμα που με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξεταστεί τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια. Είναι σε θέση αυτά τα όσα απαιτούνται να τα υλοποιήσει επαρκώς και ικανοποιητικά ή όχι. Ή μετά υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, και κενά που ε, διαπιστώνονται. Αυτό ήθελα από πλευρά αρχής εκ προημίου να αναφέρω. Έχετε νομίζω στα χαρτιά σας και το σχέδιο γνωμοδότησης για τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή το δικό μου σχέδιο γνωμοδότησης. Λέω λοιπόν για, γενικά για την αξιολόγηση όσον αφορά σφάλματα και ελλείψεις από το ελεκτικό συνέδριο πρέπει να διαφοροποιήσουμε κάπως τα πράγματα σε αυτό. Υπάρχουν διαφορά. Υπάρχει διαφορά αν υπάρχουν προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν υπάρχει κοινή διαχείριση Επιτροπής Κρατών Μελών και ιδιαίτερα που υπάρχουν προγράμματα στον εξωτερικό τομέα που ίσως με άλλο πύχη, με άλλο γνώμονα μετρώνται και σταθμίζονται από τη διαφορετικά προγράμματα. Υπάρχει λοιπόν διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την πρόκληση, τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όταν για παράδειγμα δούμε και στα εδάφια 2 και 3 το έχω εντάξει αυτό, αν δούμε τι συμβαίνει στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων τότε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου βρίσκει κανείς. Και για παράδειγμα στο θέμα ενός προγράμματος ανάπτυξης και που δεν βρίσκεται τόσο μακριά αυτή η χώρα που ε, έχουμε συνδράμει, διαπιστώνεται για αυτό το πρόγραμμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ έχει, υπάρχουν χρεώσεις ενώ δεν υπάρχουν τεκμήρια ότι πράγματι έγιναν αυτές οι πληρωμές και δαπανήθηκαν με τον ε, ενδεδειγμένο τρόπο. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, έχει μεγάλη εμβέλεια. Δηλαδή οι δαπάνες πρέπει με βάση αποδείξεις ε, να γίνονται και όχι με κατεκτήμηση υποθέσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δαπανών έχει προβλέψει την επανόρθωση, την ε, ε, επιστροφή στη σωστή τάξη πραγμάτων αυτού του θέματος. Είναι σημαντικό όταν πρόκειται για προγράμματα εξωτερικού πεδίου που πρέπει να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε. Για το θέμα των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών δεν θα πω τίποτα. Προσδοκώ και αδειμονώ να ακούσω τις παρατηρήσεις του εκπροσώπου του ελεγκτικού συνεδρίου όταν προσέλθει. Πιστεύω ότι σε αυτά τα τρία-τέσσερα κέντρα βάρους πρέπει να επικεντρωθούμε. Αφενός δηλαδή στο θέμα των εξωτερικών σχέσεων, των προγραμμάτων στην εξωτερική βοήθεια και τα ποσοστά σφάλματος ε, που διαπιστώνονται και το θέμα των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών και, τι, και εκείνα που άλλοτε είχαμε συζητήσει ποια συνέχεια θα πρέπει να δίνεται με την ανεξάρτητη αξιολόγηση από πλευράς των δράσεων αυτών ε, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στους χιώδεις εισηγητές. Από τους σοσιαλδημοκράτες. Υπάρχει κάποιος. Uh, uh, Εν γέννη συμφωνούμε με τη θέση του εισηγητή. Πολλές λογικές προτάσεις. Το μόνο που μας ενοχλεί είναι αυτή η μανία που έχει το ΕΛΚ στην παράγραφο 7 με τα business centers στην Ασία. Εμείς ε, τα θεωρούμε, θεωρούμε ότι κάνουν καλή δουλειά, προωθούν τη γνώση και την ε, ε, διαδίδουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το επιχείρημα πέραν του προπολογισμού είναι ότι θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να τα πάνε καλύτερα, αυτό θα ισχύει για τα μεγάλα κράτη-μέλη, ενώ τα μικρότερα ε, θα χάσουν αν δεν υπάρχει παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ε, παρουσία των business centers στην Ασία. Κατά τα άλλα θεωρούμε ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τον εισηγητή και έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Ευχαριστώ κύριο Κάμπαλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετική, εντυπωσιακή έκθεση. Συμφωνούμε με την απογοήτευση του εισηγητή ότι υπήρχε ουσιώδες επίπεδο σφάλματος σε όλες τις πληρωμές. Είναι περίεργο που παραμένει τόσο υψηλό και θα πρέπει να φροντίσουμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δουλειά της και να επιβάλλει την σωστή, σωστή, το έλεγχο των δαπανών και όχι μόνο εντός της Επιτροπής αλλά και στα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε περίοδο λιτότητος όταν κράτη-μέλη καταβάλουν τόσο μεγάλη προσπάθεια να περιορίσουν το κόστος. Επίσης εντυπωσιαζόμαστε, μας σοκάρει το γεγονός ότι το 89% των συναλλαγών που ελέγχθηκαν στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων ε, βοήθειας είχαν σφάλμα σε επίπεδο 29% και αυτά δεν ε, διαπιστώθηκαν από τους ελέγχους της Επιτροπής. Άρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί δεν διαπιστώθηκαν αυτά τα σφάλματα και εάν θα εγκαταστήσουν ελέγχους ώστε να εξασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν. Τέλος, όσον αφορά αφορά τη μελέτη αντικτύπου. Δεν θεωρούμε ότι, υπάρχει, ότι έχει δοθεί επαρκής προσοχή στην μελέτη αντικτύπου των εμπορικών συμφωνιών, που για μας είναι σημαντική, σημαντικό για το μέλλον. Ευχαριστούμε, Μαρίκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για το σχέδιο γνωμοδότησης που θίγει πολλά σημαντικά ζητήματα διαπιστώνουμε ότι το περιθώριο σφάλματος για τις εξωτερικές σχέσεις και τη διεύρυνση είναι σχετικά περιορισμένο, αλλά υπάρχει ε, περιορισμό, ε, περιθώριο για βελτίωση. Είχαμε στο παρελθόν μεγαλύτερα σφάλματα, η εξαφάνιση βοήθεια στην Αίγυπτο και θέματα της υπηρεσία εξωτερικής βοήθειας. Υπάρχουν ε, περιθώρια βελτίωσης και ενώ τα προβλήματα αυτά πρέπει να βελτιωθούν στα πλαίσια της ΑΦΕΤ και της ΣΥΝΤΑ, υπάρχει και άλλη επικάλυψη. Παλαιότερα έχουμε συζητήσει για την ανάγκη ενός καλύτερου συντονισμού των εξωτερικών σχέσεων και του εμπορίου ως μέρους των εξωτερικών σχέσεων. Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις εμπορικές συμφωνίες που θα συζητηθεί ευρύτερα νομίζω σήμερα, δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο σημαντικής βελτίωσης και στο χώρο της μελέτης αντικτύπου, αλλά και για την εκτονιστέρων των ελέγχους και πιστεύουμε ότι οι προτάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου θα ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, δεν είναι μόνο δημοσιονομικό το θέμα, αλλά στην ουσία πρέπει να τηρηθούν ε, οι δεσμεύσει των εταίρων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, περιβαλλοντικών προτύπων κλπ. Έτσι λοιπόν συνολικά ο έλεγχος θα δώσει καλύτερη εξοπιστία και αποτελεσματικότερο από ε, προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την κατάθεση αυτού του σχεδίου έκθεσης που συνολικά μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Τρία, τρεις παρατηρήσεις θα είχα όμως. Θέλω να τονίσω τρία πράγματα. Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ότι γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιο βαθμό οι πληρωμές αυτές γίνονται με ικανοποιητικό τρόπο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σαφέστερο τρόπο να αποσαφηνίζει πράγματα και τα ποσοστά σφάλματος όχι μόνο να τα αποκαλύπτει, αλλά να βλέπει πώς συνέβησαν και γιατί αυτά. Και συμφωνώ όσον αφορά τις επιπτώσεις με τους συναδέρφους εκ των υστέρων να δούμε τι συμβαίνει, όχι μόνο για την χρηματοοικονομική διάσταση, αλλά να δούμε όλες τις επιπτώσεις που υπάρχουν στα επιμέρους κεφάλαια μέσω τέτοιων συμφωνιών για παράδειγμα. Όλες αυτές οι πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και αυτό έχει πραγματικές επιπτώσεις στις πληρωμές, ιδιαίτερα όσον αφορά την, ε, την πτυχή της ε, βοήθειας. Θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή κατά πόσον κάποιες ε, πτυχές όχι μόνο στην εξωτερική εμπορική πλευρά αλλά και όσον αφορά και την εξωτερική πολιτική καλύπτονται. Πρέπει να είμαστε σαφέστατοι σε σχέση με τα εμπορικά θέματα. Να πούμε, να αναφερόμαστε στα μέσα τα οποία παρακολουθούμε και ελέγχουμε ως Επιτροπή για αυτές τις πτυχές. Κατά τούτο λοιπόν μια αποσαφήνιση γιατί δεν επαρκούν για μένα, δεν είναι επαρκή η σαφήνεια των, σημείο, των σημείων 1 και 2. Στο σημείο 4 κατεπίγουσα ανάγκη είναι σε σχέση με τη δράση μας ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή στο νέο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τώρα στο δεύτερο ημίση, στο τέλο του 2014, όπου πολλές νομικές πράξεις έχουν ε, ε, περάσει για την μακροοικονομική βοήθεια μελλοντικά να μην χρειάζεται πάλι να ξανακερδίσουμε το δικαίωμα των, του να θέτουμε ερωτήσεις και να διατυπώνουμε παρατηρήσεις να μην υπάρχει δηλαδή ένας ραγδαίος ρυθμός που δεν επαρκεί ώστε να κάνουμε τη σωστή δουλειά. Στην επόμενη έκθεση διαφορετικά του ελεγκτικού συνεδρίου θα δούμε σημεία και τέρατα αν δεν δράσουμε σωστά. Και πρέπει νομίζω να και τον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και Ουκρανίας να τον εξετάσουμε προσεκτικά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Οι σκιώδεις των πρασίνων δεν παρίστανται εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Κυρία Λεπέν, δύο λόγια για την έκθεση αυτή. Αναφερθήκαμε ήδη στον αριθμό σφαλμάτων που μας παρουσιάστηκε σαν κάτι στο οποίο πρέπει να υπομένουμε. Αλλά από το ηλεκτρικό συνεδρίο μαθαίνουμε ότι υπάρχουν ε, πολλά απλήρωτα στον προϋπολογισμό το 2014 φτάνουμε στα 30 εκατομμύρια απλήρωτα. Δηλαδή, όπως φαίνεται, δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τιμολόγια που δεν μπορεί να πληρώσει, να εξοφλήσει. Δηλαδή, χρεώνεται, το οποίο έρχεται σε αντίφαση με τις συνθήκες. Και θέλω να κάνω μια απληρώτηση πώς μπορούμε να δίνουμε μαθήματα δημοσιονομικά σε διάφορες χώρες και στη Γαλλία, στη χώρα μου, όταν δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε σωστά τα οικονομικά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί τους κανόνες των δικών της συνθήκων, συσσωρεύει χρέη και ανεξόφλητα ε, χρέη και όπως φαίνεται η λιτότητα ε, παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές. Ευχαριστώ από την Επιτροπή. Ο κύριος Πίτερ Σέντλερ, παρακαλώ. And, uh, thank you Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την γνωμοδότηση αλλά και για τις παρατηρήσεις του. Θα απαντήσω εν συντομία σε τρία από τα σημεία που έθεσε. Πρώτον, το θέμα του ποσοστού σφάλματος και των πληρωμών συνεχίζει να αποτελεί σοβαρό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ως τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ε, ε, πρόσφατα επισημάνθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, έχουμε δώσει έμφαση στο να ενισχυθεί μια στάση ενίσχυσης των επιδόσεων ε, και θα εφαρμόσουμε και θα παρακολουθούμε τις διαδικασίες του προϋπολογισμού όπως και τις δαπάνες. Βεβαίως η απαλλαγή είναι κάτι το οποίο το προωθούν και τα μέσα ενημέρωσης κάθε χρόνο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι κάθε ευρώ δαπανάται αποτελεσματικά και πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Το πρόβλημα με τα ποσοστά ασφάλματος μας ε, ανησυχεί στον τομέα των εξωτερικών ε, σχέσεων υπάρχει μια μειωτική, πτωτική τάση σε σχέση με το 2012 στους τομείς που παρακολουθεί η δική σας επιτροπή και το, το σχόλιο του κυρίου Σόλτς ε, είναι χαμηλό το ποσοστό και δεν εντοπίστηκαν στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου τα ποσοστά σφάλματος. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα στο δείγμα τους. Τώρα, ένα σχόλιο σε σχέση με τα business center, με τα επιχειρηματικά κέντρα. Θεωρώ ότι το μήνυμα που υπάρχει είναι ότι η Κομισιόν όπου διατηρεί τα business center αυτά έχει έναν χρήσιμο ρόλο συμπληρωματικό των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμπλέκεται απευθεία στην πρόθεση του εμπορίου, όμως το κέντρο στο Πεκίνο ε, είναι πολύ αποτελεσματικό στη δουλειά του, εξασφαλίζει ότι υπάρχει μία ευρωπαϊκή φωνή για να ασχολείται με θέματα πρόσβασης στην αγορά και εμποδίων που υπάρχουν στην αγορά της Κίνας. Είναι σημαντικό, αυτό που είναι σημαντικό στην συνέχιση ύπαρξη αυτών των κέντρων είναι να δημιουργούνται και να λειτουργούν με τρόπο που να συνάδει με το τοπικό περιβάλλον. Όταν δημιουργούνται νέα κέντρα είναι σημαντικό να αξιολογείται ο αντίκτυπός τους και η δυνατότητα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα. Το τελευταίο μου σχόλιο δεν είναι σχόλιο αφού θα επανέλθει και το ελεκτικό συνέδριο που ψιάζουμε σε κάποια από αυτά τα ζητήματα για τη μελέτη αντικτύπου και την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτή τη φάση θέλω απλώς να πω ότι το θέμα αυτό το αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εξηγήσουμε μετά την ομιλία του ελεγκτικού συνεδρίου, ποια βήματα έχουν λεφθεί. Θεωρούμε ότι βελτιώνεται συνεχώς η ανάλυση μας, αλλά βεβαίως μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής μας κύριος έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ πρώτα για την πρόταση. David, δεν έχουμε αιμονές όσον αφορά τα ε, επιχειρησιακά κέντρα, business centers. Αλλά και εμείς θα έπρεπε να ενδιαφερόμαστε να έχουμε μια αξιολόγηση για πιστοποίηση και πιστοποίησεις και τα λοιπά. Και ίσως μπορούμε να πετύχουμε μια σωστή λύση. Το θέμα της διαφοροποίησης όσον αφορά τα αίτια για διάφορα τμήματα του προϋπολογισμού που έχουμε διαφορετικά θετικές εξελίξεις σε αυτά, μπορούμε έτσι να το προσεγγίσουμε. Και το θέμα της μακροοικονομικής βοήθειας. Συμφωνώ με τα όσα είπατε. Γενικά, από πλευράς ελέγχου του προϋπολογισμού, επί πολλά χρόνια είχαμε μεγάλες αντιπαραθέσεις και για προγράμματα όπου εμείς είμαστε οι κυριότεροι χορηγοί για δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών για παράδειγμα είχαμε μακρά μακράν παράθεση. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου δεν είχε ευκαιρία να εξετάσει το τι γινόταν σε σχέση με τέτοιες δράσεις ε, των ε, Ηνωμένων Εθνών. Όμως ε, αυτό σε αντιδιαστολή με τα κράτη-μέλη. Τόσο αξιοπερίεργες είναι κάποιες δομές όσον αφορά τα διεθνή προγράμματα. Κατά πόσον τώρα στις εξωτερικές σχέσεις η διεύρυνση της εξωτερικής βοήθειας μπορεί να εξεταστεί είναι εξειδικευμένα θέματα. Εντάξει, συμφωνώ να το δούμε, αλλά να δούμε και τι θα κάνουμε με την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ. Δηλαδή, να δούμε τις εξωτερικές πτυχές υπό το πρίσμα του εμπορίου με μεγαλύτερη ακρίβεια, πιο εξειδικευμένα. Και αφενός αυτά τα οποία έχουμε everything but arms, όλα εκτός από όπλα, στο πλαίσιο του εμπορίου, είχαμε και μια επισητιστική βοήθεια δύο δις που έπρεπε να δρομολογηθεί κατά το παρελθόν γιατί δεν είχε κονδύλια ο Οργανισμός τηνών Εθνών. Αξίζει να δει κανείς τα προγράμματα, αναπτυξιακά προγράμματα και εκτός της βοήθειας αυτής που χορηγούμε να δούμε τι, τι συμβαίνει με αυτά τα ε, προγράμματα. Αξιοπρόσεκτα και αξιοπερίεργα πράγματα συμβαίνουν πολλές φορές και πρέπει όλα αυτά να τα δούμε. Και για την σωστή ανάπτυξη της κάθε χώρας ε, να δούμε ποιες επιπτώσεις έχουν όλα αυτά στις εμπορικές πτυχές. Ε, κάτι το οποίο πριν από λίγες μέρες παρατήρησα είναι για κάθε ευρώ λέει αναπτυξιακής βοήθειας που δίνουμε σε κάποιες χώρες 10 ευρώ είναι αξιοπρόσεκτο από κάποιους διάβλους βγαίνουν από αυτή τη χώρα. Ε, πρέπει να δούμε ισχύει αυτό ή όχι. Νομίζω δεν μπορεί να ισχύει, αλλά είναι πολύ αξιοπρόσεκτα. Τέτοια πράγματα να δούμε. Δεν έχω απάντηση τώρα σε αυτό που είπατε, αλλά αποκινούμε την ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, Επιτροπή Εξωτερικών και Επιτροπή Ανάπτυξης, πρέπει να τα συζητήσουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, αυτά είναι τα θέματα και που από δική μου πλευράς την γνωμοδότηση θα ήθελα να τη συμπληρώσουμε και μετά θα δω και τις τροπολογίες σας για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά λέει ο Πρόεδρος. Η δυνατότητα να καταθέσετε τροπολογίες θα υπάρχει μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου αγαπητοί συνάδελφοι, 12 το μεσημέρι. 11 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι κατάθεση τροπολογιών ώστε στις 21-22 Ιανουαρίου στη συνεδρίασή μας να μπορούμε να ψηφίσουμε αυτές τις τροπολογίες προς έγκριση. Ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο ημερήσιας διάταξης, επανερχόμαστε στο 5 της ημερήσιας διάταξης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουμε τον κύριο Τομέ τώρα ανάμεσά μας. Καλώς ήρθατε κύριε Τομέ. Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ειδική έκθεση για τις ε, προτιμησιακές συναλλαγές, καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών ε, αναφέρθηκε και στην έκθεση έχουμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές που εμπεριέχονται που αξίζουν να εξεταστούν κάπως πιο αναλυτικά και σε μεγαλύτερο βάθος να αναλυθούν, ώστε η πολιτική μας στο μέλλον να μπορέσει να βελτιωθεί. Χαίρομαι που ο κύριος Τομέ είναι εδώ και μπορεί να μας δώσει μια εισαγωγή στα αποτελέσματα της, ε, ε, για τα αποτελέσματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχετε τον λόγο κύριε Τομέ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Πρόεδρε, με αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΙΝΤΑ, ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για τις, ε, ε, του 2014 για το κατά πόσο είναι κατάλληλη διαχείριση των καθεστώτων προμετρησιακών συναλλαγών. Χαίρομαι που παρίσταμε εδώ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για να σας παρουσιάσω προφορίες σχετικά με το έργο μας. Όπως θα γνωρίζετε, 22 Σεπτεμβρίου είχα ήδη την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Πιστεύω ότι το έγγραφο εργασίας που παρουσιάστηκε από τον κύριο Στάς αντιμετωπίζει και αναφέρεται πολύ κατάλληλα στα συμπεράσματα και τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου. Θα ξεκινήσω δίνοντας σας μια επισκόπηση του τι ήταν ο έλεγχος και τι λέει το ελεγκτικό συνεδρίο στην ειδική του έκθεση. Το ελεγκτικό συνεδρίο εκτίμησε το κατά πόσο είναι σωστή η διαχείριση των προτιμησιακών ε, συναλλαγών. Αποτελούν ένα βασικό μέσο εμπορικών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Αποφέρουν ωφέλη οικονομικά τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις εταίρες χώρες. Συνεπώ η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά για τη διασφάλιση των συμφερόντων τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αποτελούν κομμάτι τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για αρρωγή των οικονομιών ε, των τρίτων χωρών για τη βοήθεια στην εκρίζωση της φτώχειας και στην δημιουργία ανάπτυξης. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τέτοιες διευθετήσεις καλύπτουν το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 183 χωρών η αξία των αγαθών όπου εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των ε, συναλλαγών ε, αντιστοιχεί σε 242 δισεκατομμύρια ευρώ, 14% των εισαγωγών. Ήταν διτό ο στόχος ε, της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα αξιολόγησε κατά πόσο η Κομισιόν αξιολόγησε σωστά τις οικονομικές επιπτώσεις των προτιμησιακών συναλλαγών τόσο πριν από την υπογραφή όσο και μετά από τη θέση σε ισχύ τους. Δεύτερον, ο έλεγχος προσπάθησε να διαπιστώσει κατά πόσο η έλεγχη των εισαγωγών ε, τέτοιων προϊόντων ε, είναι αποτελεσματική ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν ε, υπάρχει κάποιο ανέτιο όφελος προς, ε, ε, για, την ύπαρξη χαμηλών δασμών για τέτοια προϊόντα. Τώρα θα σας πω ποια ήταν τα συμπεράσματα. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, όσον αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων, των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η Κομισιόν χρησιμοποιώντας τα μέσα εκτίμησης δεν εκτίμησε όλες τις οικονομικές επιπτώσεις των συμφωνιών που έχει συνάψει. Έτσι λοιπόν, οι υπεύθυνοι χαράξεις της πολιτικής και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι δεν ενημερώνονται επαρκώς για τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις των εμπορικών διευθετήσεων. Αξιότιμα μέλη δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται τη συμφωνία TTIP με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπιστώσεις του ελεκτικού συνεδρίου έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η συμφωνία TTIP, όπως ονομάζεται, δεν έχει ελεγχθεί από το ελεκτικό συνέδριο, διότι τη στιγμή που έγινε η εκτίμηση, η εκτίμηση αντικτύπου δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί. Ελπίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα λάβει υπόψη τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου και θα αξιολογήσει οικονομικά όλες οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης σχετίζεται με τους ελέγχους που διενεργούνται επί των ε, εισαχθέντων αγαθών. Ε, Γεννούνται σε τρία επίπεδα αυτή η ελέγχη. Πρώτον, εφαρμόζεται από τι τελωνιακές αρχέ των κρατών μελών. Δεύτερον, γίνονται έλεγχοι στις ε, εταιρούς χώρες και τρίτον επίβλεψη της Κομισιόν. Ο έλεγχος εστιάστηκε στα συστήματα ελέγχου που έχουν εγκαθιδρύσει τα κράτη-μέλη αφενός και στην επίβλεψη της Κομισιόν αφετέρου. Από αυτή την άποψη το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι τα κράτη οι τελεινικέ αρχές των κρατών μέλων θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι μόνο ε, κάποια συγκεκριμένα είδη ωφελούνται των ε, μειωμένων δασμών, αλλά διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Και δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα ε, βρίσκεται στον πίνακα 4 της έκθεσης, όπου αναφέρεται σε μια περίπτωση εισαγωγής σκόρδο από το Μεξικό, με προτιμησιακούς δασμούς, ωστόσο όμως το σκόρδο αυτό προερχόταν από την Κίνα και συνεπώς δεν ήταν επιλέξιμο για προτιμησιακή μεταχείριση. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίε στους θελωνιακούς ελέγχους που εφαρμοζόνται από τις αρχές ορισμένων ε, κρατών μελών που ελέγχθηκαν. Σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εισαχθέντων προϊόντων που ελέγχθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο σε πέντε κράτη-μέλη, διαπιστώθηκε ότι πολύ συχνά τα έγγραφα που τεκμηρίωναν ε, την προτιμησιακή αντιμετώπιση έλειπαν σχετίζονταν με εισαγωγές του 2009 και δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν οικονομικά διότι έχει παρέλθει η τρίτη περίοδος. Και έτσι λοιπόν τα αντίστοιχα έσοδα έχουν χαθεί. Το ελεγκτικό συνέδριο εκτίμησε ότι η απώλεια ανερχέται σε 655 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί σε 6% των τελωνιακών δασμών της υποελεγχό ε, χώρας. Παρόμοια προβλήματα διαπιστώθηκαν στο δείγμα των εισαγών του 2011, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι εθνικές τελωνιακές αρχές έχουν ακόμα χρόνο να επιβαλούν ε, οικονομικές διορθώσεις και να εφαρμόσουν τις διαπιστώσεις του ελεκτικού συνεδρίου σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα από τους αγωγές. Είναι πως εκεί δεν έγινε κάποιος υπολογισμός της απώλειας. Επίσης διαπίστωσε ο έλεγχος ελλείψης στην επίβλεψη της Κομισιόν στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Κατά την άποψη του Ελεγχτικού συνεδρίου, οι σημερινές ε, νομικές διατάξεις των ε, προτιμησιακών διευθετήσεων δεν περιλαμβάνουν αρκετές εγγυήσεις για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αξιότιμα Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, το ελεγκτικό συνέδριο εξέδωσε μια σειρά συστάσεων μετά από αυτές τις διαπιστώσεις ώστε να βελτιωθεί η αξιολόγηση των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών. Το ελεκτικό συνέδριο λοιπόν θεωρεί ότι η Κομισιόν πρέπει να διεξάγει σε βάθος ολοκληρωμένη και ποσοτικοποιημένη ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων κάθε νέας συμφωνίας ε, προτιμησιακών συναλλαγών και για αυτό το σκοπό η Κομισιόν θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του εμπορίου θα πρέπει να λαμβάνουν όλες τις σχετικές αναλύσεις έγκαιρα. και τα στοιχεία της Eurostat ε, για την ποιοτική αξιολόγηση. Επίσης η Κομισιόν θα πρέπει να διεξάγει εξ post αξιολογήσεις, εκ των υστέρων αξιολογήσεις, ώστε να εκτιμά το βαθμό στον οποίο οι προτιμησιακές ρυθμίσεις ε, εκπληρούν τους ε, στόχους πολιτικής και πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η απόδοση σε τομεί κλειδιά. Για να αυξηθεί η προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν θα πρέπει να δημιουργήσει προφίλ Eurex, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο των αναλύσεων για τη μείωση των ε, ε, διαφυγόντων εσόδων από τον προπολογισμό της Ένωσης. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου ρίξου. Πρέπει επίσης ε, να γίνονται επισκέψεις παρακολούθησης βάσει επικινδυνότητας σε χώρες εξαγωγών που εποφελούνται από προτιμησιακή μεταχείριση για να αποφύγονται απώλειες ε, εσόδων ε, λόγω παρέλευσης ε, των προθεσμιών θα πρέπει η Κομισιόν βασίζεται και σε έρευνες της Όλαφ και να ενισχύσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αμοιβέ εμπορικές διευθετήσεις και να χρησιμοποιεί περισσότερο τις αρχές προφυλάξης και διασφάλισης. Τέλος, το ελεγκτικό συνέδριο θεωρεί ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προωθήσει την αντικατάσταση των πιστοποιητικών που υπάρχουν τώρα με πιστοποιητικά των εξαγωγέων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ja, ganz Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Τομέ. Πολύ προσεκτικά παρακολούθησα όσα μας είπατε. Και συμβαίνει το ίδιο όπως όταν διάβασα για πρώτη φορά την έκθεσή σας Είπα στην αρχή, για κοίτα, έκανε μια έκθεση πάλι εδώ το Ευρωπαϊκό ε, Ελεκτικό Συνέδριο, πολύ ωραία. Όταν τη διάβασα όμως ε, με ηλέκτρισε, διότι τα όσα αναφερόντουσαν, θεμελιώδη ερωτήματα για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διατυπώνουν, ερωτηματικά θέτουν. Και όταν συνειδητοποιεί κανείς αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή ανεπαρκής εξ άντε ή εξ αναλύσεις για την ταυτοποίηση του τι συμβαίνει και οι πληροφορίες που στοχεύουν σε μάσα ε, να μην είναι επαρκείς δηλαδή το ότι εμείς ε, για την επαρκή ενημέρωση για τα μειονεκτήματα και προτερήματα και για τις επιπτώσεις και για το αν μια συμφωνία εμπορίου επιτυγχάνει αυτά που επιθυμούμε ή όχι με κάνει και ανησυχώ πολύ αν δεν βελτιωθούν όλα αυτά αυτές οι ανεπάρκειες και αυτά τα κενά πώς μπορούμε να συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες και να προχωρούμε. Έχουμε 20 διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή για τέτοιες συμφωνίες. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φυσικά. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε αυτά τα κακό κείμενα να επανορθωθούν. Ακριβώς για την TTIP, τη συμφωνία με τις ίπα εμπορίου και επενδύσεων. Τι κάνει ώστε να υπάρχουν στοιχεία αξιόπιστα στη διάθεσή μας. Ακριβώς όταν έχουμε μια πολύ φιλόδοξη ημερήσια διάταξη και την δίκανη σε αυτή για όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις στο χρονορίζοντα που έχουμε. Πρέπει πραγματικά αξιόπιστες πληροφορίες να δίνονται και όχι με κενά και με λήψεις. Αυτά για να τονίσω το πόσο με εμπλέκει αυτό το θέμα και με συγκλώνησε. Ο κύριος Μπέγκε, εισηγητής, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά την περίληψη την ξαναδιάβασα, έριξα μια ματιά και καθίσατε σαφές ότι αφενός υποστηρίζω αυτό που είπατε, Πρόεδρε έχουμε ένα πολύ περίπλοκο σύνθετο πεδίο ενώπιόν μας. Πρόσφατα είχα πάει στο Αμβούργο και είδα το λιμάνι του Αμβούργου και τον τεράστιο αριθμό εμπορευματοκιβωτίων, κοντέινερ και σκέφτηκα ποιος θα τα ελέγχει και πώς όλα αυτά. Είναι πραγματικά ε, μια, μια παραφροσύνη και ταυτόχρονα το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε μια πολύ σκόπιμη και εύθετη ανάλυση των ε, πραγμάτων. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε αυτό. Ερώτηση προς το, προς το ελεγκτικό συνέδριο. Ποια, βρίσκουν, ποια είναι τα ευάλωτα σημεία, τα ευαίσθητα σημεία. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπάρξουν προφίλ χαρακτηριστικά κινδύνων. Υπάρχουν λήψεις ε, στην ε, επαγρύπνηση όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει. Δηλαδή πόσα στελέχη χρειάζονται για να τα βγάλει πέρα η Επιτροπή με αυτή τη δουλειά για να γίνονται, γίνονται σωστά τα πράγματα. Ή μήπως εδώ υπάρχουν διαφοροποιημένες προσεγγίσεις για τα ουσιοδέστερα πιο ευάλωτα σημεία όσον αφορά την υλοποίησή τους από τα κράτη-μέλη. Σημεία τα οποία αναφέρθηκαν που κατά το ίμιση είναι σημεία που αφορούν τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως. Και το ενδιαφέρον ερώτημα είναι πού να ξεκινήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φυσικά εκείνη που δίνει την υποστήριξη και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση αυτών των μέτρων των κρατών μελών και πρέπει επιτόπου να γίνεται ο έλεγχος. Ευχαριστώ. Εσείς έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια <clears throat> κύριε Τόμε και στο ελεγκτικό συνέδριο για αυτό το έργο. Διότι πιστεύω όπως κατέδειξε ο κύριος Τομέ, είναι μια μελέτη αποτελεσματική περιεκτική για τα ποια θέματα μπορεί να δημιουργούν προβλήματα στην εμπορική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για μένα όπως είπε ο Πρόεδρος, με ανησύχησε αυτή η έκθεση. Με ανησύχησε πρώτα απ' όλα για την έλλειψη στοιχείων και ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια σειρά θεμάτων. Και αυτό δεν είναι εντάξει, πρέπει να επανορθωθεί, να διορθωθεί. Διαπραγματευόμαστε πολλές συμφωνίες εμπορίου που είναι πολύ σημαντικές αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας. Και επίσης βλέποντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις της ε, επαρκούς και εξαντλητικού ελέγχου. Βέβαια είναι δύσκολο όλα τα, όλα τα πάντα να ελέγχονται, και τα κράτη-μέλη και έναντι των κρατών μελών. Πρέπει να υπάρξει αυστηρότητα έναντι αυτού του θέματος. Πιστεύω πραγματικά στο ελεύθερο εμπόριο, αλλά με ίσες ευκαιρίες και με ισότιμο πλαίσιο για όλους. Πρέπει να είναι σεβαστοί οι κανόνες. Διαφορετικά δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται οι συμφωνίες εμπορίου για, ως πόρτα και παράθυρο για να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με παράνομο τρόπο. Και υπάρχουν και επιφυλάξεις από πλευράς πολλών Ευρωπαίων σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες ελευθέρων, ελεύθερου εμπορίου. Και υπάρχουν και οικονομικές δυσκολίες για τους Ευρωπαίους. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτά τα θέματα για να μην υπάρξει ευκαιρία να ε, παρακάμπτονται και να υπονομεύονται αυτές οι διατάξεις. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί λοιπόν. Αυτό που θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη, να τα προτρέψει, να υλοποιήσει τα, τις, ε, τα απαιτούμενα, τα προαπαιτούμενα. Να κάνει και ίδια το ίδιο. Να επαγρυπνούμε, τουλάχιστον να διασφαλιστούν οι εγγυήσεις τι συμβαίνει και να έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε και να τα επανορθώσουμε αν χρειαστεί. Ε, σε ευχαριστώ από τους σοσιαλδημοκράτες, ο Ντέιβιντ ή ποιος. υποθέτω ότι θέλω να σχολιάσω τρία ζητήματα. Πρώτον, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο από αυτή την έκθεση είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι νομικές δυνατότητες να αντιμετωπιστεί η απάτη σε τρίτες χώρες. Όταν κάνουμε ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου δεν έχουμε κατά ανάγκη μια συμφωνία με τους εταίρους που να μας επιτρέπει να δράσουμε από αυτού. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε στις επόμενες ε, συμφωνίες, αμοιβές ε, συμφωνίες, ώστε όταν αντιμετωπίζεται απάτη να υπάρχει δυνατότητα ο εταίρος να υποχρεωθεί να δράσει από αυτής. Δεύτερον, ίσως δεν κατάλαβα τα επιχειρηματά σας εδώ, αλλά αυτό το πιστοποιητικό προέλευσης είναι αυτοπιστοποίηση. Θα βελτιώσει αυτά τα πράγματα. Εγώ θα θεωρούσα ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε ακόμα περισσότερο την απάτη για τον εξαγωγέα. Γι' αυτό θα ήθελα να με εξηγήσετε τη λογική της προτασίας που είμαι βέβαιος ότι υπάρχει. Ε, αυτό που είπατε κι εσείς και ο πρόεδρος με έκανε να σκεφτώ ότι δεν είστε πεπισμένοι από τους εκ των ε, αξιολογήσεις για την απώλεια εσόδων. Όπως και σε πολλούς άλλους χώρους, ας πούμε λέμε ότι αν αλλάξουμε την υποστήριξη στα γεωργικά προϊόντα ή την κατάρτιση υπάρχει απώλεια ε, εσόδων στα κράτη-μέλη. Εμείς δεν ζητάμε να γίνει μια ανάλυση των εσόδων που προέρχονται από αυτές τις εξαγωγές. Ε, τα έσοδα που χάνονται στις εμπορικές συμφωνίες είναι δύσκολο να καθοριστούν, γιατί όπως γνωρίζετε, καμιά φορά το εμπόριο πηγαίνει αλλού, οπότε κάποιοι άλλοι χάνουν ή κερδίζουν λόγω της αλλαγής των δασμών, αυξάνει το εμπόριο, άρα το ε, το απολυστέν έσοδο δεν είναι ολόκληρο αυτό το οποίο υπολογίζεται. Άρα αυτό το που είπε ο Χέλμουντ Σούλς σε άσχετο θέμα προηγουμένως είναι ε, ουσιαστικό, δηλαδή η εκ των υστέρων ανάλυση θα πρέπει να ενδιαφέρεται για το ποιο είναι τα ωφέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις χώρες αποδέκτες, τι έχει γίνει για την κοινωνική πολιτική και για το περιβάλλον. Γιατί το να επικεντρωθούμε μόνο στα έσοδα δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Ευχαριστώ κύριε Σκέπρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι συντομία σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν επί του 6, μάλλον τα είπα στο 6 αλλά επιπλέον. Αυτό μας ε, ανησυχεί σε σχέση με τις πιθανές οικονομικές απώλειες με από τα σφάλματα αυτά. Μοιάζει ότι τα ποσά είναι σοβαρά και λόγω της οικονομικής κατάστασης, ε, ιδιαιτέρως ε, λόγω αυτής, θα πρέπει να τους δοθεί προτεραιότητα. Και δεύτερον, είναι σημαντικό το προσωπικό να να προσπαθεί να βρει ποιοτικά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε καλύτερη ανάλυση από πλευράς Eurostat επίσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίκε. Από τη μία πλευρά μας δίνει νέα στοιχεία που πρέπει να σκεφτούμε. Από την άλλη πλευρά επιβεβαιώνονται πολλά που είχαμε πει στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε ένα ε, πεδίο ίσο για όλους όπου θα, υπάρχουν, θα υπάρχει επιβολή, αξιολόγηση, εκτίμηση, να μην υπάρχουν κενά ώστε οι χώρες να μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς. Νομίζω έχει μεγάλη σημασία να γίνονται ανεξάρτητες εκτιμήσεις, έλεγχοι και να επιβάλλεται να επιβάλλονται οι κανόνες, πρέπει να υπάρχουν συγκριτικοί δείκτες που θα ε, επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανέρχεται, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος που θα μπορεί να παίξει το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας, για να μπορέσουμε να ζητήσουμε ευθύνε από τους υπευθύνους. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ντέιβιτ Μάρτιν για την απάτη. Είναι πολύ ανησυχητικό. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ ανέφερα την έκθεση του δικαστηρίου για την Αίγυπτο στο παρελθόν. Ήταν αδύνατο να διαπιστώσουμε αν τηρήθηκαν οι συγκριτικοί δείκτες, γιατί πρώτον δεν ήταν σαφείς και δεύτερον υπήρξαν πάρα πολλέ περιπτώσεις όπου πλέον τα χρήματα δεν μπορούσαμε να τα εντοπίσουμε. Δεν ξέρουμε πού ήταν. Ίσως πήγαν σε καλό σκοπό, ίσω όχι. Αλλά αυτή η αβεβαιότητα και η δυνατότητα που υπάρχει για απάτη και κατάχρηση από άλλε χώρε είναι πάρα πολύ σοβαρή ώστε να την αποδεχτούμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ενισχύσουμε του μηχανισμού ελέγχου, την δημοκρατική επιτήρηση και να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές ε, ελέγχου ώστε να είναι πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όσα κάνει. Τόσο και για τις προ... προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες αλλά και ευρύτερα. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν φαντάζομαι να επεκταθούν και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ. Πράγματι, ευχαριστώ Χέλμουντ. Ευχαριστώ Μπέρντ για αυτές τις παρατηρήσεις με τις οποίες συμφωνώ είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητη η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Και όταν τίθεται το θέμα για την εμπορική μας πολιτική με αυτά τα ερωτήματα, μπορώ να πω ότι συμφωνώ τώρα. Γιατί? Γιατί αφορά τους δύο νομοθέτες ουσιαστικά και που είναι υπεύθυνοι και αποφασίζουν για τη χρήση κονδυλίων των φορολογουμένων. Και δεν θέλω εμείς να ευθυνόμαστε εμείς για την κατάσταση μεταξύ των κρατών μελών και για τις νομικές προϋποθέσεις έχουμε το νομικό καθήκον εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ελέγξουμε επακριβώς τι γίνεται με την χρήση αυτών των κονδυλίων. Και γι' αυτό το ερώτημα, το οποίο ίσως προς τον εισηγητή και προς τον κύριο Τομέ του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν θα ήταν αναγκαίο εμείς για κάθε νομοθετικό έργο, πράξη νομοθετική, για κάθε συμφωνία να έχουμε μια τέτοια αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποβάλλει τέτοιου είδους στοιχεία για αξιολόγηση που έναντι πραγματογνωμοσύνης μπορεί κανείς να δει τι γίνεται και για τα ερωτήματα τα οποία και ζητήματα που τίθενται να ξέρουμε τι γίνεται σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, αυτές τα, αυτά τα θέματα. Και για τα κράτη-μέλη συγκεκριμένη υποχρέωση να αναλαμβάνεται στο κρατικό επίπεδο να ασκείται πλήρως ε, η ευθύνη ελέγχου. Δηλαδή να προβληματιστούμε γι' αυτό, να δούμε πώς μπορούμε στην υλοποίηση του έργου ελέγχου οι συμφωνίες αυτές όσον αφορά τα κράτη-μέλη να μπορούν να εντάσσονται σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή η, κρατικές, η κρατική ευθύνη να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που επομίζονται και αναλαμβάνουν τα κράτη. Να προβληματιστούμε και να δούμε πώς κάτι τέτοιο μπορεί να διαμορφωθεί αποτελεσματικά σε μια τέτοια κατεύθυνση να πορευθούμε ιδιαίτερα όσον αφορά και τις, ε, την ε, δράση του ελεκτικού συνεδρίου. Πράγματι, και αυτό είναι το έργο μας θα έλεγα, τις συνέπειες αυτές ε, να τις παρακολουθήσουμε. Τι λέει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά. Τι λέτε, αδειμονώ να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Τόμε. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Δεν θα σας κάνει έκπληξη που η Κομισιόν πιστεύει τα εξή. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεχόμαστε την έκθεση και τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Θεωρήσαμε ότι η διαδικασία αυτή ήταν εξαιρετικά χρήσιμη μας βοηθάει να προσαρμόσουμε τον τρόπο εργασίας μας όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και όσον αφορά και τη τελωνιακά θέματα, ε, τα, τις τελωνιακές διαδικασίες στα κράτη-μέλη. Σημειώνουμε τις διαπιστώσεις του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ελεκτικό συνεδρίο έκανε μια αξιολόγηση για ένα διάστημα 15 ετών. Και το ίδιο το ελεκτικό συνεδρίο αναγνωρίζει ότι άλλαξε μορφή η μελέτη μέσα στο διάστημα αυτό, άλλαξαν μορφή οι αξιολογήσεις. Ε, αν δούμε λοιπόν τη σημερινή κατάσταση, οι εμπορικές μας συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών με την Ιαπωνία και την TTIP, ε, που βέβαια δεν εντασσόταν στο πεδίο αυτού του ελέγχου, υπόκεινται σε ανάλυση σε τέσσερα στάδια ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάνουμε την εκτίμηση που πριν ξεκινήσουν. Κάνουμε μία αξιολόγηση βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ε, Διανεργούμε μια ανάλυση στο τέλος των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τις επιπτώσεις των συμφωνιών πριν έρθει για υπογραφή στο Συμβούλιο και για επικύρωση στο Κοινοβούλιο. Και επίσης ε, κάνουμε, και αυτό είναι ε, σίγουρα κάτι το, για το οποίο το ελεκτικό συνέδριο επισήμενε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ε, κάνουμε εκ των υστέρων αξιολογήσεις ώστε να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα σε διάφορους τομείς των συμφωνιών που έχουμε συνάψει. Αυτό σχετίζεται και με τα όσα ανέφερε ο David Μάρτιν. Ένα από τα πράγματα που επισημαίνει το Ελεκτικό συνέδριο είναι τα απολεσθέντα έσοδα. Αυτό προσπαθεί να το αξιολογήσει στην εκτίμηση αντικτύπου της Οικομισιόν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι κάτι που μελετάμε στι αξιολογήσει εκ των υστέρων, στι εξπόστα αξιολογήσει. Αλλά δεν είναι αυτή όλη η ιστορία. Φυσικά όταν υπάρχει μια εμπορική συμφωνία, ένα από του σκοπού είναι η μείωση των δασμών και στην μείωση των εσόδων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως... ελπίζοντα ότι οι συναλλαγέ μα θα γίνουν πιο ανταγωνιστικέ, θα δημιουργήσουν θέσει εργασία. Φυσικά είναι σημαντικό να μετρηθεί αυτό ο συγκεκριμένο δείκτη, αλλά ε, το θέμα δεν αφορά μόνο τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο θέμα φυσικά είναι ότι αναγνωρίζουμε πως στο παρελθόν κάποιες από τις αξιολογήσεις που κάνουμε κάποιες από τις εκτιμήσεις αντικτύπου θα μπορούσαν να ήταν πιο αξιόπιστες και πιο ολοκληρωμένες. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή επικαιροποιούμε τις εσωτερικές, εσωτερικές γραμμέ γραμμές ε, για τις εκτιμήσεις ε, ε, βιωσιμότητας. Έχουμε το έργο του ελεκτικού συνεδρίου, Έχουμε συμφωνήσει, έχουμε κάνει μια νέα συμφωνία με τη Eurostat για να εμπλέκονται πολύ περισσότερο, πολύ πιο στενά στην ε, επαλήθευση των δεδομένων που χρησιμοποιούμε εμείς για τα οικονομικά μας μοντέλα. Επίσης ε, σημειώσαμε ότι κάποιος από τους τομείς ε, που διαπιστώθηκε από το συνέδριο ότι δεν είμαστε τόσο αξιόπιστοι όσο θα έπρεπε είναι, αφορούν συγκεκριμένου τομεί. Για παράδειγμα, στην Ινδία επέκριναν το γεγονό ότι δεν καταφέραμε να μετρήσουμε, να αξιολογήσουμε τι επιπτώσει στην αεφορία ε, σε θέματα ε, άτυπης οικονομίας, ε, μαύρης οικονομίας. Εμείς έχουμε δυσκολία να αξιολογήσουμε αυτή την οικονομία ακόμη και στα δικά μας κράτη. Σε μια άλλη περίπτωση για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μας επέκριναν γιατί δεν συμπεριλάβαμε αξιολόγηση των ζητημάτων πρόσβασης σε φάρμακα. Πολύ συγκεκριμένος τομέας και συμφωνώ, ναι, αν δεν καλύπτεται δεν μπορεί κανείς να πει ότι η ανάλυση είναι ολοκληρωμένη. Από την άλλη όμως, ε, θεωρούμε ότι σήμερα η ανάλυση είναι ικανοποιητική. Χρησιμοποιούμε ένα αξιόπιστο μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέω ε, ε, ως οικονομικό μοντέλο. Έχουμε μία αξιολόγηση ευρεία επιπτώσεων ε, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε, πριν οριστικοποιήσουμε αυτές τις μελέτες. Όσον αφορά τις αξιολογήσει εκ των υστέρων, όπω είπα, δεχόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και το έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε τρεις αξιολογήσει ex post για το επόμενο έτος, Πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο έτος είναι φυσικά σημαντικό να αφήσουμε αρκετό χρόνο ώστε να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των συμφωνιών. Πολλές συμφωνίες δεν φέρνουν επιπτώσεις μέχρι ε, μετά από πενταετία. Χρειάζεται κάποιες διατάξεις να τεθούν σε ισχύ. Η πλήρης επιπτώσεις, τα πλήρη αποτελέσματα δεν είναι αίσθητα ένα, δύο, τρία χρόνια μετά από την πρώτη θέση σε ισχύ, ε, ή μάλλον προσαρμογή, ε, συγγνώμη, προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Πολλές φορές χρειάζεται να αφήσουμε χρόνο. Και τέλος, να αναφερθώ στο σημείο που ακούσαμε για το κατά πόσο υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι και νομικοί έλεγχοι των εμπορικών μας συμφωνιών. Ε, αυτό που συζητήσαμε πιο συγκεκριμένα με το ελεγκτικό συνέδριο είναι κατά πόσο πρέπει να εντάξουμε στις εμπορικές μας συμφωνίες το ενδεχόμενο αναστολής της ε, εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων σε θέματα τελωνιακής συνεργασίας με τις αρχές μια τρίτη χώρα. Η συζήτηση αυτή ανακύψε ουσιαστικά διότι όταν ξεκίνησε ε, η διαδικασία έλεγχου δεν είχε περάσει πολύ καιρό μετά από τη συμφωνία. Ε, πρότεινε λοιπόν η Κομισιόν μια τέτοια διάταξη αναστολής και σε μια συμφωνία, τη συμφωνία με την Κορέα, δεν μπορέσαμε να αποσπάσουμε τέτοιου είδους δέσμευση από τους Κορεάτες. Και τελικά ω διαπραγματευτέ, χρειάστηκε να λάβουμε μια απόφαση για την όλη ισορροπία τη διευθέτηση. Ε, μας έδωσαν κάτι άλλο, αλλά το μηχανισμό που αφορά τη διαβούλευση με του κορεάτε πριν από την αναστολή. Μα έδωσαν αυτό, δηλαδή μπορεί να γίνει αναστολή, αλλά όχι τόσο εύκολα όσο αν ήταν μονομερή ο μηχανισμό αναστολή. Σε επακολούθε, σε επόμενε συμφωνίε όπως με τη Σιγκαπούρη και τον Καναδά, που σύντομα θα έρθουν εδώ στο Κοινοβούλιο, θα δείτε ότι αυτή η διάταξη έχει συμφωνηθεί. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε δεσμευτεί. Και μεριμνομώστε να είναι κομμάτι του βασικού πακέτου διαπραγματευσής μας. Χωρί να επηρεάζει τις καλές μας σχέσεις με την τρίτη χώρα. Το τρίτο που θέλω να πω σχετίζεται με κάποια ζητήματα τελωνιακά. Θα ήθελα να επισημάνω το ζήτημα που αναφέρθηκε του risk profiling, του προφίλ επικινδυνότητας. Και αυτό γίνεται τώρα από τη Γενική Διεύθυνση Τάξου. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένους τομείς υψηλή επικινδυνότητας και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να ε, επιστήσουμε την προσοχή τους σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, συγκεκριμένους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα λάθος εφαρμογής των κανόνων. Η ουσία είναι ότι δεχόμαστε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θεωρούμε ότι είναι μια υποφιλής άσκηση που μας βοηθά να βελτιώσουμε περισσότερο τη δική μας, τις δικές μας μέθοδους ανάλυσης. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, διότι εν τέλει, αν δεν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι συνάπτουμε συμφωνίες με βαρύ βάση που επιτυγχάνουν τα αποτελέσματά τους, και αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχουν παρασχεθεί αυτά τα αποτελέσματα μέσω αξιολογήσεων ex τότε γυρνάμε σε αυτά που είπατε στην αρχή, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε μια ουσιώδη έλλειψη εμπιστοσύνη ε, στο... στις... σε όλε τι εμπορικέ μα ε, διαδικασίε. Ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μα βοηθήσει η έκθεση αυτή. Ο θέλει να λάβει τον λόγο και πάλι, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Κάπως όταν είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι κάποια πράγματα ήταν ε, ε, στην ώρα τους, άλλα πράγματα μετά από πέντε χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια δεν θα είναι το ίμιση από εμάς εδώ παρόν. Και γι' αυτό αυτό μετάραξε που άκουσα και γι' αυτό η πρόταση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει έγκαιρα να τύχει συνέχεια. Το θέμα δηλαδή των χαρακτηριστικών κινδύνου που πρέπει να εκπονήσουμε δηλαδή να ξεκινήσουμε αναφέρθηκε τουλάχιστον και να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνων και συστημάτων κινδύνου τα κράτη-μέλη. Να μην πάνε χαμένε οι προσπάθειες και οι συστάσεις της έκθεσης. Και οι χώρες ε, που θα τύχουν αυτής της προτιμησιακής βοήθειας και να γίνουν διακριβώσεις επιτόπου και να δούμε και σε σχέση με τους κανόνες προέλευσης τι μπορεί να γίνει. Αυτά είναι οι πυρήνες, ε, τα ουσιοδέστερα στοιχεία των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει μια ενδιάμεση έκθεση που θα λέει ποια είναι η τάξη η κατάσταση πραγμάτων μετά από αυτή την πρώτη διακρύβωση και να μας πει μήπως είναι θετική εξέλιξη ή είναι, ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Να τα δούμε αυτά και μετά να μπορέσουμε να δράσουμε και να δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστώ. Äh, Κύριε και εγώ έτσι ακριβώς το βλέπω πως εσείς. Ίσως λοιπόν να μπορέσουμε να συντάξουμε μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαριθμούνται αυτά τα στοιχεία και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να δώσουμε συνέχεια και να έχουμε και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα καταθέσουμε για αυτό το θέμα. Βλέπω συγκατανεύεται, συμφωνείτε να το κάνουμε λοιπόν. Ας συντάξουμε αυτή την κοινή επιστολή προς την Επίτροπο και να υπάρξει follow-up, συνέχεια που θα δοθεί σε αυτό το θέμα. Κύριε Τομέ, Έχετε κάποιες ερωτήσεις λοιπόν που σας δόθηκαν, ακούσατε τις απόψεις της ε, Επιτροπής, είναι η σειρά σας τώρα να τοποθετηθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν απαντήσεις τις οποίες θέλω να δώσω, όμως προηγουμένως να υπογραμμίσω ότι η έκθεσή μας δεν ε, ουδόλως αμφισβητεί την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μελετήσει κάποιες κρίσιμες πλευρές όπως είναι η ενημέρωση που διατίθεται για την διαδικασία διαπραγματεύσεων και έχουμε κάνει συστάσεις για την βελτίωση των, της κατάστασης. Δεν αμφισβητούμε την εμπορική πολιτική βοηθούμε τη βελτίωσή της. Αυτό προσπαθούμε με, την, με τις εκθέσεις μας. Με τα χαράς μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πλέον είναι έτοιμοι να αποδεχτούν κάποιες από τις συστάσεις μας και σε μερικά χρόνια θα ε, παρουσιάσουμε την επόμενη έκθεσή μας και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε εδώ ώστε να εξηγήσουμε πώς κατά τη γνώμη μας ε, έχουν ληφθεί υπόψη οι συστάσεις μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε, πράγματι έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις αδυναμίες παρά στα ωφέλη της εμπορικής πολιτικής. Αυτός ήταν ε, ο σκοπός και της έκθεσής μας, να κάνουμε συστάσεις ε, για βελτίωση. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, οι νομικές ε, δυνατότητες, οι νομικές εξουσίες των εμπορικών ρυθμίσεων. Εν γέννη η Όλαφ έχει δυνατότητες να κάνει έρευνες. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν μπορεί να το κάνει ε, σε τρίτες χώρες και σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες έχουμε κάνει αναφορά η, εφαρμογή ε, των συστάσεων της Όλαφ από τις τελωνιακές αρχές έπρεπε με κάποιο τρόπο να εγκριθούν από την ε, χώρα εξαγωγής. Αυτές είναι οι αλλαγές που συνιστούμε. Αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις, όμως το θέμα αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση. Υπάρχει και το θέμα της αυτοπιστοποίησης. Και πάλι ε, αυτό σημαίνει ότι οι εισαγωγείς αναλαμβάνουν την ευθύνη. Οπότε οι εισαγωγείς οι οποίοι εποφελούνται από πιστοποιητικά προέλευσης μπορούν να κάνουν επίκληση στην ε, καλή πίστη. Οπότε αναλαμβάνουν την ευθύνη. σε κάποιους τομείς ε, φορολόγησης. Ε, η αυτοπιστοποίηση συνεπάγεται ε, αλλαγή στον αριθμό των ανθρώπων. Δεν συνιστούμε να αυξηθούν οι τελωνιακοί. Εμάς μας απασχολεί το θέμα της αποτελεσματικής συνεργασίας και της επατελεσματικής παρακολούθησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεσή μας αναφέρονται περιπτώσεις όπου οι συστάσεις της Όλαφ δεν έγιναν δεχτές από τις εθνικές αρχές ή δεν λήφθησαν υπόψη από τις εθνικές αρχές και η διοικητική συνεργασία κρατών μελών δεν λειτουργήσε ε, αποτελεσματικά. Δεν ζητάμε περισσότερους ανθρώπινους ή υλικούς πόρους επιδιώκουμε την καλύτερη αντιμετώπιση των συστάσεων, την καλύτερη διαχείριση των συστάσεων. Τα περισσότερα από τα θέματα που θίγουμε και τα περισσότερα από τα θέματα που προκύπτουν από τις μελέτες αντικτύπου είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Εμείς δεν μπορέσαμε να ε, μετρήσουμε τον αντίκτυπο, αλλά θέλουμε να δούμε πώς, ποιες είναι οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε, αυτά τα σχετικά νέα μέσα που, έχουμε στη, που υπάρχουν στη διάθεσή μας, τα θεωρούμε ε, βελτίωση υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει τέτοιου είδους αναλύσεις με τρόπο συνεπή σε κατάλληλο χρόνο. Είναι κατάλληλες αυτές, είναι σωστές αν δεν γίνουν πολύ καθυστερημένα και, να και, αν δεν και αν στηρίζονται σε δεδομένα. Φυσικά Υπάρχουν ανησυχίες για το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο όμως αυτή τη στιγμή είναι κατά πάσα πιθανότητα το βέλτιστο διαθέσιμο εργαλείο. πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα δεδομένα θα έχουν επικαιροποιηθεί όταν ε, εισάγονται στο μοντέλο, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Μερικά άλλα ζητήματα. Οι πιθανές οικονομικές απώλειες. Είπαμε ότι έχουμε ποσοτικοποιήσει συγκεκριμένα στην έκθεσή μας. Προηγουμένως, στο θέμα της απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφερθήκατε στα σφάλματα. Εδώ διαπιστώσαμε ότι στις χώρες που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκαν σφάλματα στον τομέα των εσόδων, ουσιώδη και ε, σημαντικά. 6% των συνολικών τελωνιακών εσόδων. Αν δείτε τον ε, προπολογισμό εσόδων, δεν είναι μεγάλο το ποσό, παρά τα αυτά είναι 152 εκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο. Είναι ουσιώδες από, μόνο από δύο κράτη-μέλη. Ε, όπως αναφέρεται στην έκθεση, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Γαλλία. Όλοι πρέπει να γίνουν, να δουλέψουν πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Σε όλες οι τελωνιακές αρχές πρέπει να κάνουν πολλά. Με ρώτησαν αν θεωρεί το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, ότι πρέπει να ε, όλες οι διαδικασίες να υπόκεινται σε αυτή την ε, ε, ρύθμιση. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δικαιολογείται η μελέτη αντικτύπου. Οι περιστάσεις λόγω του επίγοντος της συμφωνίας συνεπάγεται ότι δεν μπορούν να γίνονται πάντοτε εκ των προτέρων μελέτες αντικτύπου, αλλά αυτό πρέπει να έχει δικαιολογηθεί από γνωμοδότηση της Επιτροπής. Βεβαίως υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα, η δυνατότητα του εκ των υστέρων ελέγχου, της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Θεωρούμε ότι τρία χρόνια μετά την θέση ενισχύ της συμφωνίας είναι επαρκής χρόνος για μια ενδιάμεση αξιολόγηση που θα είναι χρήσιμη στους, ε, σε αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν για την πολιτική και για να μπορέσει να αξιολογηθεί η συμφωνία. Νομίζω ότι απάντησα στα θέματα που τέθηκαν, σχεδόν σε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Μπορούμε να σας απαντήσουμε γραπτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε, όπως και οι απαντήσεις που δώσατε, όπως συμφωνήσαμε. Προηγουμένως θα στείλουμε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρακολουθήσουμε τις συστάσεις σας με προσοχή και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε σε άλλη συνεδρία της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Χαίρετε. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt. Εντάξει, αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στην κοινή συζήτηση που είναι το σημείο 7 και το σημείο 8 και που είναι <clears throat> για την αναδιατύπωση δύο νομοθετικών προτάσεων για τις εισαγωγές, ιδιαίτερα προς το προϊόντων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ουσιαστικά είχαμε σχεδιάσει μέσα στο πλαίσιο της συζήτησης για τα κλωστοϊφαντουργικά και την κατάσταση στο Μπαγκλαντές να εξετάζαμε. Διότι παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τι γίνεται με τις βελτιώσεις των όρων εργασίας και διαβίωσης ε, των ε, εργαζομένων γυναικών και ανδρών στο Μπαγκλαντές μετά από εκείνο το φοβερό ατύχημα την πυρκαγιά. Ο, πυρ, ο πρέσβης όμως του Μπαγκλαντές δεν ήταν σήμερα διαθέσιμος, δεν μπορούσε να προσέλθει. Και έτσι στην επόμενη συνεδρίασή μας του Ιανουαρίου θα συζητηθεί το θέμα του Μπαγκλαντές. Έχουμε τις δύο νομοθετικές προτάσεις τώρα. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Βαλένσα, εισηγητής για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, τα σχέδια εκθέσεων μου είναι έτοιμα. Η ουσία της πρότασης της Κομισιόν είναι σε μεγάλο βαθμό τεχνική. Πρόκειται λοιπόν για τεχνικές διορθώσεις λαθών ε, που διαγράφηκαν. Πρώτα απ' όλα στον πιο γενικό κανονισμό που αφορά τις εισαγωγές εκτός κλωστοϊφαντοργικών προϊόντων. Η κύρια αλλαγή αφορά την αφαίρεση ορισμένων χωρών από το πράρτημα επειδή πλέον είναι μέλη του ΠΟΕ. Αρμενία, Ρωσία, Τατζικιστάν και Βιετνάμ. Αυτές είναι οι χώρες που είναι πλέον μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται τώρα η καλύψη της πρότασης σε εισαγωγές από Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Βόρεια Κορέα, ε, Τουρκμενιστάν και Ουσμπεκιστάν. Δεύτερον, όσον αφορά την πρόταση για τις εισαγωγές υφαντουργικών προϊόντων, η προηγούμενη διαδικασία λήψη αποφάσεων του άρθρου 23 αντικαταστάθηκε από απόφαση υπό τη διαδικασία εξέταση όπως συμφωνήθηκε υπό την Omnibus 1. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο τομέα τη κλωστοϊφαντουργία είναι πολύ ευαίσθητο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή οι μόνε χώρε από τι οποίε εισάγει υφάσματα κλωστοϊφαντουργικά ήδη η Ευρώπη και που δεν καλύπτονται από πρωτόκολλα ή άλλε συμφωνίε είναι η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα. Ο κανονισμός ε, ορίζει ετήσια ποσοτικά όρια για τις εισαγωγές κλωστοφοδορικών προϊόντων από αυτές τις δύο χώρες και επιτρέπει την εγκαθίδρυση μέτρων επίβλεψης ε, και επίσης τέτοια μέτρα προβλέπονται για εισαγωγές κλωστοφοδορικών προϊόντων από άλλες τρίτες χώρες που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Όπως ανέφερα στην προηγούμενη συνάντηση, οι δύο αυτές προτάσεις κωδικοποιούν υπάρχοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κοινών κανόνων που αφορούν την επίβλεψη και τα μέτρα επίβλεψης και ε, προστασίας ε, σε θέματα τέτοιων εισαγωγών. Η παγίωση λοιπόν, ε, η ενοποίηση αυτών των ε, τροπολογιών ε, καθιστά τις προτάσεις πιο φιλικές προς το χρήστη είναι τεχνικές και δεν αποτελούν το αντικείμενο διαφορών. Υπάρχει όμως μια παράληψη σε αυτή την πρόταση αναδιατύπωση για τις εισαγωγές κλωστοφαδρικών προϊόντων που εγώ παρατήρησα και εντόπισα και χρειάζεται διόρθωση. Αναφέρομαι στο άρθρο 9.2 της αναδιατυπωμένης έκθεσης ε, ε, κατάλογος θεσμικών οργανών και αξιωματούχοι που πρέπει να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Αυτό παρατήρησα εγώ, διότι δεν αναφερόμαστε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ θεσμικών οργάνων και να οδηγήσει σε αποκλεισμό του Κοινοβουλίου. Μια παρόμοια διάταξη περί εμπιστευτικότητας απορρίτων πληροφοριών υπάρχει και σε άλλες αναδιατυπωμένες προτάσεις που δεν αφορούν τα κλαστοϊφαντουργικά και στην άλλη πρόταση, στο άρθρο 5.2, αλλά εκεί δεν αναφέρεται ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο στον κατάλογο. Επειδή ο αρχικός κανονισμός εισαγωγής κλωστοφεντρικών προϊόντων ε, είναι του 1994, ε, ίσως αυτός να είναι ο λόγος, επειδή είναι τόσο παλιός. Θα μπορούσε η Γενική Διεθνή Εμπορίου να μας εξηγήσει γιατί το Κοινοβούλιο δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 9.2. Και επίσης το Συμβούλιο προτείνει μια σειρά τροποποιήσεων ε, στην αναδιατύπωση ε, τη, του κανονισμού για το κλασιτοφοδρικά προϊόντα. Φαίνονται τεχνικής φύσης, αλλά θα μπορούσε να μας εξηγήσει η Προεδρία τι αφορούν και πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαλέσα. Τώρα από τους σοσιαλιστές, ε, Αλέσια. Ναι, ευχαριστώ. Επειδή οι αναδιατυπώσεις αυτές είναι τεχνικής φύσης, ε, δεν έχω ιδιαίτερα πράγματα να προσθέσω. Ωστόσο, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία γενικότερα για να υπογραμμίσω κάτι που σκέφτηκα μετά το τελευταίο που είπε ο κ. Συσίγητης, δηλαδή το ρόλο του Κοινοβουλίου, το νέο ρόλο του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Και συνεπώς ε, να τονίσω την αναγκαιότητα ότι και αυτοί οι κανονισμοί πρέπει να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα πιο εντατικής ε, ανταλλαγής και πιο συχνής ανταλλαγής ε, απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων ε, και πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί επίβλεψης σε περίπτωση ενεργοποίησης μηχανισμών επίβλεψης σε κρίσιμες καταστάσεις. Θυμόμαστε ότι σε ορισμένες χώρες υπάρχει υπερβολική, υπερβολικό πλεόνασμα ε, overcapacity για κάποιους τομείς ε, σημαντικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέμβουμε και το Κοινοβούλιο να έχει στα χέρια του όλα τα στοιχεία ώστε να μπορέσει να ασκήσει πίεση σε περίπτωση που απαιτείται τέτοια παρέμβαση. Το αναφέρουμε αυτό και σε σχέση με μια πιο ευρία ανησυχία αφορά μια τάση που εμείς διακρίνουμε αυτή τη στιγμή σε ορισμένες ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες τάσεις προστατευτισμούς ειδικότερα σε ορισμένους τομείς και αυτές οι τάσεις δεν ευθυγραμμίζονται με τη νέα φάση εμπορικής πολιτικής που εμείς ξεκινάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό έδειξε και η συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτός ο κανονισμός και η ραδιατύπωση αυτών των κανονισμών παρότι τεχνικές αυτές οι ραδιατυπώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευκαιρία για να επισημάνουμε το θεσμικό ρόλο του Κοινοβουλίου ε, και το ρόλο των ε, διοργανικών σχέσεων με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Και μετά η ΣΥΑΣ. Ανταλούν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ με τον εισηγητή. Ε, ε, ε, έχω υποβάλει από τις 5 Νοεμβρίου κάποιες ερωτήσεις και από τις απαντήσεις προκύπτει ότι τα μέτρα αυτά ε, προστασίας σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Είναι ενδιαφέρον που ε, διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, να είναι στη διάθεσή μας. Είναι πολύ χρήσιμο για χώρες όπως η Βόρεια Κορέα. Είναι χρήσιμο όταν ξέρουμε για ποια προϊόντα πρόκειται. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας όπως είπε και ο εισηγητής. Φυσικά Θέλουμε να επιμείνουμε στην ε, σημασία. Όπως είπε ο εισηγητής, τα θέματα είναι εξαιρετικά τεχνικά. Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις, όμως προσυπογράφουμε ε, τα ερωτήματα που έθεσε ο εισηγητής. Εν γέννη συμμεριζόμαστε τις απόψεις των κρατών μελών και τις νομικές υπηρεσίας ε, που θεωρούν ότι τα θέματα είναι εξαιρετικά τεχνητικά. Ευχαριστώ. Μαρίκε. Thank you, Chair. Uh, thanks. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά του. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Συμφωνούμε με τα θέματα που καλύφθηκαν και με την πρόταση και την προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρη, διαφανής και να παρέχει νομική ασφάλεια η νομοθεσία. Και άρα ε, δεν θα προτείνουμε οποιαδήποτε τροπολογία, δεδομένου ότι αυτά υπάρχουν στο κείμενο. ο Χέλμουτ, ευχαριστώ πάντα Να ζητήσω συγγνώμη που δεν παρίσταται η σκιώδηση η συγγήτριά μας. Με παρακάλεσε να αναφέρω ότι στις τεχνικές προσαρμογές ε, για τις οποίες, ε, ε, τις οποίες εξετάζουμε μια παρατήρηση από την ομάδα μας σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή που ευχαριστώ γι' αυτό και που νομίζω ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα των όγκων, των ποσοτήτων και των παρατημάτων αλλά και για τους όρους Πώς δηλαδή επιτόπου παράγονται τα κλωστοϊφαντουργικά επιτόπου, τους όρους και προϋποθέσεις παραγωγής τους. Αυτή η πτυχή στα σκεπτικά, στο σκεπτικό, στα, ε, επιχειρήματα ή στα εδάφια να μπορέσει να ενταχθεί. Δηλαδή ζητείτε ώστε οι νέες αλλαγές που θα υπάρξουν ευθύς εξ αρχές να ληφθούν υπόψη τα ζητήματα αυτά που θα πρέπει να ενταχθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και θα λάβει τώρα η Επιτροπή τον λόγο για να τοποθετηθεί. Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Μαριάννα Κνασέσκου παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Τη σημείωσα. Θα αναφερθώ σε μια συγκεκριμένη παρατήρηση που αφορά την πολύ αυτή τεχνική, την εξαιρετικά τεχνική αυτή υπόθεση. Πράγματι, στην Omnibus, στον κανονισμό των διασφαλίσεων, η αναφορά στο Συμβούλιο έχει απαλληφθεί. Γιατί το Συμβούλιο δεν θα εμπλέκεται πλέον στην εφαρμογή του κανονισμού, εμπλέκεται η επιτροπολογία. Δεν έχουμε εντοπίσει το ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, ε, έχει απαλληφθεί από τον κανονισμό των κλειστιφαντουργικών και επισημαίνουμε και ε, χαιρόμαστε για το ε, σφάλμα αυτό που επεσήμανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τροπολογία επ' αυτού, εμείς ε, θα την αποδεχτούμε. Όπως είπα προηγουμένως, σημειώσαμε τις παρατηρήσεις σας για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα τις έχουμε κατά νου στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Με, με τα χαράς θα μελετήσω καλύτερα τις προτάσεις Προεδρίας. Ως εισηγητής θα φροντίσω να εξασφαλιστούν τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά από όσα άκουσα προλίγου, θα ήταν νομίζω σωστό να υποβληθεί τροπολογία ώστε να... Ε, σε σχέση με το Συμβούλιο στο άρθρο 9.2. Επίσης ε, θα διαγραφεί το Συμβούλιο στο 9.2 και θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις Προεδρίας. Αλλά επειδή όμως και τα δύο, οι δύο αυτοί φάκελοι είναι τεχνικοί και καθόλου αμφιλεγόμενοι, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμφωνία. Δηλαδή να επέλθει συμφωνία πριν από την επίσημη πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Και ελπίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής θα συμφωνήσουν με την άποψή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οπότε, τροπολογία, ε, ημερομηνία υποβολη τροπολογιών, 15 Δεκεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Η συζήτηση θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, 21 Ιανουαρίου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε τώρα μένει κάποιος χρόνος μέχρι τις 11, οπότε θα αρχίσει και η συνεδρίαση των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Ευχαριστώ πολύ.